Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνεδρίαση. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω. Έχουμε μια ολόμεστη ε, ημερήσια διάταξη και θα πρέπει να κάνουμε όσο δυνατόν γρήγορα τη δουλειά μας. Ξεκινάω λοιπόν πολύ πολύ γρήγορα. Η μερίσια διάταξη αν τη δέχεστε όπως την έχουμε προτείνει. Έχει κάνει αντιρρήσεις. Ουχή. Και εγκρίνεται. Όσο Σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Ε, διερμηνία έχουμε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, πορτογαλικά, ουγγρικά, πολωνικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και σας υπενθυμίζω ότι η παρούσα συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Η συνεδρίαση των 22 Ιανουαρίου είναι τα συμπεράσματα στη θέσή σας. Σας απεστάλθη σαν στις 24 με το email και εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις θεωρείται ότι έχουν εγκρίθει που δεν αγγέλθησαν να μέχρι τις 26 Ιανουαρίου. Έχουμε πολλούς, ε, πολλά πληρεξούσια για την ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία και καλό και τους εισηγητές, τα και εισηγητρίες, όσο το δυνατόν να αποφύγουν τις ε, τοποθετήσεις πριν από τις ψηφοφορίες. Υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις παράλληλα πολλών συναδέλφων μας, γι' αυτό καλό θα ήταν να προχωρήσουμε γρήγορα για να τους αποδεσμεύσουμε. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe, Κυκλοφορία για την προσωπική συμφωνία από τη διοργανική διαπραγμάτευση. Ξέρετε ότι έχει να κάνει αυτό με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων. Έχω, ο συνάδελφος κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει εξασφαλίσει, η συνάδελφος κυρία Κώστα έχει εξασφαλίσει τη συμφωνία. Παρακαλώ πολύ σύντομα, ναι, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Κάναμε καλή δουλειά, πιστεύω, με μια καλή συμφωνία που τηρεί ακριβώς και τις απαιτήσει και διεκδικήσεις της δικής μας Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη δουλειά, λέει η Πρόεδρος, και προχωρούμε στην ψηφοφορία. Μία και μόνη προσωρινή συμφωνία ηλεκτρονικά και έρχεται. Ich schließe die Abstimmung. «24 υπέρ, 2 κατά και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Και έτσι προχωρούμε με την πρόταση αυτή στην Ολομέλεια και περνώ σε μια μακροσκελή ψηφοφορία στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι η πρόταση για μια νομοθετική έκθεση της κυρίας Helga Trippel για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Helga Trippel, θέλεις να πεις κάτι, παρακαλώ, στα αγγλικά. Καλημέρα συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομη. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία για το θέμα αυτό. Όλοι σχεδόν είμαστε πεπισμένοι ότι είναι καλό να προχωρήσουμε προς πεστορία αλληλεγγύη και δυνατότητες ε, για εθελοντική εργασία για τους νέους και κυρίως τους πιο, σε αυτούς που βρίσκονται σε πιο δύσκολες ε, συνθήκες, όχι δηλαδή για τους προνομιούχους, δυνατότητες για ε, ανάπτυξη κοινωνικών δυσμών και κοινωνική ενσωμάτωση, μια νέα κοινωνική προσέγγιση για το πρόγραμμα αυτό που πιστεύω ότι θα αποδειχθεί όπω και το Erasmus Plus, ε, ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο στόχο ο δικό μα και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον. Ε, νομίζω ότι είναι καλό να αλλάξουμε τον τίτλο ωστόσο, γιατί ο όρος σώμα, ε, θελοντικό σώμα ή σώμα εθελοντών δεν ακούγεται πολύ καλά σε αρκετές γλώσσες, γι' αυτό θα προτιμούσα να πούμε σώμα και, εθελοντών και αλληλεγγύης. Περισσότερα πράγματα λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, αλλά επειδή δεν προβλέπονται νέοι πόροι, θα πρέπει είτε να διατεθούν, ε, επειδή δεν αρκούν οι πόροι, θα πρέπει να διατεθούν νέοι, είτε θα πρέπει να βρεθούν από τα περιθώρια του, από τα αποθεματικά του πολιτισμού οικονομικού πλαισίου. Υπάρχει μια επεξηγηματική παρατήρηση η οποία με βρίσκει αντίθετη ότι δεν είμαστε εξοπλισμένοι για να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά μπορούμε με αυτήν την λύση να βοηθήσουμε στην ενσωμάτωση. Όλοι οι φορείς με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει έχουν μια σαφή εικόνα και άρα πρέπει να αλλάξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον προϋπολογισμό, όχι 80-20, απασχόληση και θελοντική εργασία, αλλά να μειωθεί, γιατί δεν είμαστε κατά των δυνατοτήτων για ανάληψη δραστηριότητας της ε, ε, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αλλά να πούμε ιδιαίτερα ότι ο στόχος μας είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στην θα αμφισβητήσουν την εντολή Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνεση, τα επιχειρήματά μας είναι καλά, είναι στεναρά και νομίζω ότι μπορούμε να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ Ελγα, για τη δουλειά. Τεράστιο το έργο, πολλές συμβαστικέ συμβαστικές που χρειάστηκε να ε, σχηματίσεις, να καταρτήσεις. Έχουμε και τις τροπολογίες της Επιτροπής ΕΜΠΛ οι οποίε στο βαθμό που υπάγονται, όπως ορίζει άλλωστε και ο κανονισμός του άρθρου 54, στις αποκλειστικέ αρμοδιότητε τη ΕΜΠΛ, ενσωματώνονται αυτομάτως στο κείμενο και δεν ε, ψηφίζονται. Προχωρώ λοιπόν στην ψηφοφορία. Στον μακροσκελή αυτό κατάλογο με την ε, τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 23, συμβαστική 23, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική 12, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 324, γυρνάμε μερικές σελίδες, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και στην 325 τώρα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 13 Α, όχι, με συγχωρείτε, 327. Με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος, 327 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται, ε, απερίφθη. Και πάμε τώρα στην 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 326 υπέρ όχι διορθώνει πρόεδρος με συγχωρείτε και εγώ τα έχω μπερδέψει συμβαστική 13 θα τα βολέψω με σύντο χρόνο θα τα πάμε καλύτερα 13 λοιπόν συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 362 εξήντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 371 γυρίσαμε μερικές σελίδες 371 Υπερκατά. αποχές απερίφθη η 46 έχει αποσυρθεί 375 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Μα τα είπα. Μα τα είπα. Λοιπόν, κάποια δυσκολία είχαμε στη ερμηνεία. 375, έτσι. Ωραία. 372 και 373 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 374 κατά πίπτη, προφορική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 376 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 35 της έμπλη υπέρ. Πρώτο τμήμα της έμπλη 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 384 και 385 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 387 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Επαληθεύουμε λοιπόν. Και άρχεται. 387 πάντα. Πέρας. 12 υπέρ, 15 κατά περίφθη. 48 υπέρ, κατά, αποχές. Έχει απορριφθεί νομίζω, αλλά να σηκώνετε παρακαλώ τα χέρια, αλλιώς δεν μπορώ να βλέπω. Επαληθεύουμε λοιπόν την 48. Πέρασε. Εγκρίνεται 14 υπέρ 13 κατά. 388. 389. Μαζί υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 390 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 της απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Απερίφθη. Α, όχι, είναι no vote. Ωραία, 18 υπέρ, κατά, από αποχές εγκρίνεται 398 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 399 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 400 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 συμβαστική α όχι, όχι συμβαστική απλώς τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 411 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 54, 412, 418 ταυτόσημες υπέρ κατά άποχες εγκρίνονται 413 υπέρ κατά αποχές Ας το επαληθεύσουμε παρακαλώ 413 Πέρας. Απερίφθη 16 ψήφοι κατά, 11 ψήφοι υπέρ. 414 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ δεν είναι σεφές το αποτέλεσμα. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ. Πέρας. 17 ψήφοι κατά, εννέα υπέρ, απερίφθη. 415 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 416 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 417 μαζί με τη ρέγγι 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 8 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 της γεωργικής υπέρ κατά αποχές να υποθέσω ότι έχει εγκριθεί αλλά στο επαληθεύσουμε «23 της Άγκρη». Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 9 κατά, εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 427 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 428 υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε, γιατί και έτσι αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. Σαράντα της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 ένα της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Temple 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 είναι χωρίς ψηφοφορία και έτσι προχωρώ 400, στην 44 της Ρέτζη υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. 44 της Επιτροπής των Περιφερειακών Υποθέσεων. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. 13 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. 431 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 433 υπέρ, κατά. 433 υπέρ, Κατά. Αποχές απεριφθεί. 434-435 χωρίς ψηφοφορία. 436-439 ταυτόσιμες, Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 437-438 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 440 υπέρ. Κατά αποχές απεριφθεί. NV21 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 26 της άγκρη υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 444 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 446 και Ρέτζι 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 445 έμπλη 43 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 22 της ένβη υπέρ κατά αποχές απερίφθη 447 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 448 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 449 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 450 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 451 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 16α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 463 463, NV23, Ρέγγι 48, ταυτός μας και οι τρεις υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Έμπλ 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 466-467 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απερίφθησαν συγγνώμη διορθώνει ο μιλήτρια απερίφθησαν ...469 υπέρ κατά. Απόχες απερίφθη, 470 υπέρ κατά. Αποχές. Απερίφθη 21 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69. 69 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 483 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 484 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 385 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 486 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 387 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλη 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 490 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 491 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβη 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην Ρέγγι 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 πεσύρθη 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτζ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 496 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 497 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 498 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 499 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 500 και NV26 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 501-502 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 503 απεσύρθη, badge 10 όχι, 504 με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μαζί με την 505, 506, badge 11, έμπλη 49 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 507 υπέρ, 508, 9 και badge 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 510 11, 12, μπάτς 13 υπέρ. Κατά Κατά, εγκρίνονται. 5, 13, 14, 15, μπάτς 14, έμπλη 50. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Έμπλη 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μπάτς 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην 520 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλη 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρη 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Μπορεί να μην είδα σωστά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Είχατε δίκιο. Είχα κάνει λάθος εγκρίνεται. Μπάτς 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 521 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβη 27. Παρακαλώ. Ένβη 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 56 υπέρ, κατά αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά παρακαλώ για να είμαστε βέβαιοι άρχιτη ψηφοφορία πέρας μεγάλη διαφορά εγκρίνεται σας παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας για να βλέπω Άγκρι 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέγγι 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 525 όχι αποσύρθη 526 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 547 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 548. Απεσύρθη. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπάτζ 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένβι 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 565 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 566 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 567 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 απεσύρθη, μπάτς 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζιτ 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 568 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 569 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να το επαληθεύσουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχιτε ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 υπέρ 14 κατά Πάτς 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 570 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 574 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 591 και 92 που ταυτίζονται υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.28. Λίγες σελίδες παρακάτω. Τη βρήκατε όλοι. 6.28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6.26. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Κανένα πρόβλημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 626. Αν θέλετε να το ξανακάνουμε με διανατάσεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 14 κατά, απορρίπτεται. 627 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 629 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 630 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Μπάτζ 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτζ 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6.36 περ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβι 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 78 υπέρ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αυτό για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε τις τροπολογίες Ρέγγι 78, ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας ψηφοφορίας, 16 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. 6.32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 απεσύρθη, 6.34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 6.39 40 41 ταυτίζονται υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Ρέτζι 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.42 6.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άγκρι 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 644, 645 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ενβι 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβη 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 649 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 650 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 651 και 656 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Έμπλη 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένβι 45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6.54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 81 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 657 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 658 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, συγγνώμη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Ρέτζι 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 659 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να το επαληθεύσουμε ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία Geschlossen. πέρας απορρίπτεται 663 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 664 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να το ξανακάνουμε. 664 υπέρ. Ναι, πράγματι, είναι διαφορετική η εικόνα τώρα. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, όχι, Πάμε στην ε, Ρέτζι 83. Ναι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 669, 670 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ρέτζι 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 673 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Envy, 46, Άγκρι 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ρέτζι 85 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνονται. 675 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 676 77, Envy 47, άγκρι 37 που ταυτίζονται. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ναι βεβαίως κανένα πρόβλημα να το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 676 έως άγκρι 37. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα, άρχιτε ψηφοφορία. Και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται 16 υπέρ 9 κατά. NV48, Άγκρι 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και περνάμε στην τροπολογία 682, nv 49, Άγκρι 39 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές,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 Εγκρίθηκε η Άγκρη 38. Περάσαμε στην 682. Όχι γιατί η 681 απεσύρθη. Λοιπόν, ξαναπάμε. 682 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV50 και 683 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Μπάτζ 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 684, 85, 86, Μπάτζ 30, ένβι 51, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και περνάμε στην τροπολογία 688, 689, 690, μπάτς 31, NV 52. Όλες μαζί από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και περνάμε στη ροπολογία 693. 94-95, Μπάντς 32, nv 53, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Άγκρι 40, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Oh, Συγγνώμη, η Άγκρη 40 καταπίπτει. Συμφορία για την τροπολογία για τις τροπολογίες 697, 698, 99, Μπάτ 33, NV 54. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνονται. Μπατ 34, NV 55, 701, 702, 703. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 705 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. εγκρίνεται. Ρέτζι 1 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. 128 υπέρ και έμπλενα 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100... Συμβαστική α. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Δεν ξέρω, καλύτερα να το επαληθεύσουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Συγγνώμη, είχατε δίκιο. Με μεγάλη διαφορά κιόλας εγκρίνεται. 24 ψήφι υπέρ, 2 κατά. Έμπλ 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170-171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Έμπλ 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. nv 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 7 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να είμαστε βέβαιοι και να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Επιστροπολογίας Άγκρι 7. Geschlossen. Mit 15 zu 12 abgelehnt. Απορρίπτεται 12 υπέρ, 15 κατά. Λοιπόν, για να δω που πάμε. Τώρα πάμε στην έμπλη 10. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 9 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά καλύτερα να είμαστε βέβαιοι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ επί της τροπολογίας Άγκρι 9 τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 13 κατά. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 221 και 222. Από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 2-2-3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ναι, weil das abgelehnt ist. 221 und 222. 2.21, 2.22 ε, απορρίφθηκαν, γι' αυτό και περνάμε στη 2-23 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Συμβιβαστική Der Kompromiss 8 war bei mir verrutscht. Συμβαστική 8. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 232. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπι 20, έμπι 19, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 240, υπέρ, κατά. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη NV6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 9α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV7 που είμαστε α υπέρ κατά αποχές απερίφθη 16 της Ρέγγι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ ρέγγι 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 254 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 46, 246 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 247 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 248 εγκρίνεται συγγνώμη 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 19 της Ρέγγι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 23 της έμπλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 της Ρέγγι υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 268 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 266 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 της έμπλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 της έμπλη και μια εγωιστική κάπως ρέγγι 23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 273 υπέρ Α, όχι, όχι. Ρέγγι 24, με συγχωρείτε. Στην προσεχή σελίδα και άγκρι 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 ρέγγι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 274 υπέρ. Κατά αποχές. Απέριφθη 275 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 270, εγκρίνεται 276 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 277 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV10 υπέρ όχι, ρέγγι 26, ρέγγι 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται άγκρι 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 281 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 282 υπέρ κατά αποχές απερίφθη NV11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 286 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 27 ρέγγι υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 287 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 291 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 288-289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 ρέγγι υπέρ κατά αποχές απερίφθη 17 άγκρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 292 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 29 ρέγγι υπέρ κατά αποχές απερίφθη 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 295 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 296 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 της ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 2 των προπολογισμών υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε 2 της Επιτροπής των Προπολογισμών Πέρας 15 υπέρ, 12 κατά εγκρίνεται. 2 των ε, προϋπολογισμών, 3 των προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές. Και νομίζω έχουμε την ίδια πλειοψηφία, αλλά στο επαληθεύσουμε. 3 της Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Πέρας. 15 υπέρ, 12 κατά. 4 των προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 299 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 5 των προπολογισμών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 30 της Επιτροπής των Περιφερειακών Υποθέσεων, Ρέγγι, 30 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 18 της Άγκρη υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 19 της Άγκρη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 26 απασχόληση έμπλ υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 300 όχι 124 124 κοντεύουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 18 υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εξαιρετική δουλειά και τώρα ψηφίζουμε την ανάθεση εντολής για διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή δυνάμει του 69C του κανονισμού μας, ηλεκτρονικά και αυτό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ονομαστική μάλιστα. Πέρας. Δεκαοχτώ υπέρ. Πέντε κατά, μία αποχή και συγχαρητήρια. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Θερμές ευχαριστίες για την υποστήριξη, για τη συγκεντρωμένη δουλειά. Έχουμε ακόμη κανένα δυο ψηφοφοριούλες. Δεν τελειώσαμε. Σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Πρόταση γνωμοδότηση για έκθεση πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμό τη ε, Οικονομική Πολιτική, Απασχόληση, Κοινωνικά, στην ετήσια έρευνα ανάπτυξης. Julie Ward, έχεις κάτι να μας πεις? Εν συντομία, θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη δουλειά τους. Ήταν καλό που μπορούσαμε να δούμε πραγματικά στοιχεία, να τα ερευνήσουμε, να δούμε τις τάσεις και να δούμε πού υπάρχει κόσμος που υπαρχει κοσμος που υστερει Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικοί, πιο περιεκτικοί, να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, στην κατάρτιση ε, για την απασχόληση στη συνέχεια. Ελπίζω λοιπόν η έκθεσή μας να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και προχωρώ στην ψηφοφορία συμβαστική παρελθόν ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 10 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 11 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13-14 υπέρ, κατά, αποχές και το επαληθεύουμε. Απερίφθη λοιπόν ένα υπέρ 16 κατά, συμβαστική 2. Δεκαεπτά υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 25 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 26 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 27 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πριν περάσουμε στην 41, ε, ε, η κυρία Σόιντροβα έχει μια προφορική τροπολογία για την οποία ενημέρωσε με email εχθέ τους συναδέλφους. Την παρακαλώ λοιπόν να μας εξηγήσει ποια είναι η προφορική τη τροπολογία, να μας την αναγνώσει και μετά να προχωρήσουμε στη δικασία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Προτείνω Αντί για πρόσφυγες να πούμε ετούνται στο άσυλο. Αντί για migrants, asylum seekers. Γιατί είναι πιο σαφές έτσι. Αυτή είναι η προφορική μου τροπολογία. Καλώς ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Προφορική τροπολογία δεν, είναι, δεν φτάνει μέχρι το σημείο του 41 που έχουμε να ψηφίσουμε τώρα. Προτείνω λοιπόν πρώτα να ψηφίσουμε το κείμενο της 41 και αν αυτό δεν γίνει δεκτό, προχωρούμε στην προφορική τροπολογία. Και έτσι ρωτώ αν έχουν αντιρρήσει συνάδελφοι για την προφορική τροπολογία. Όχι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη 41 όπως έχει. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Λοιπόν, ηλεκτρονικά την προφορική τροπολογία σας παρακαλώ. 41 αρχίζει η ψηφοφορία. Πρώτα ψηφίζουμε την 41. Πρώτα την 41 χωρίς το κείμενο. Εάν δηλαδή απορριφθεί, τότε πάμε στην προφορική τροπολογία, γιατί αυτή είναι η σωστή, αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Ψηφίζουμε την 41 μόνο, πέρας της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται και έτσι έχει, γίνει, έχει καταπέσει η προφορική τροπολογία. 38 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ και 44 μαζί υπέρ, κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 64 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρασε 13 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Πέρας. 19 υπέρ. 4 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Σημείο 6. Σχέδιο γνωμοδότηση. Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κούρτσιο Μαλτέζε. Θέλεις να λάβει το λόγο πάλι, Κούρτσιο. Θες να πεις κάτι. Ναι, πολύ σύντομα γιατί θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους, χάρη στου οποίου κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Σε ένα θέμα πολύ μεγαλύτερο, πολύ σοβαρό την εποχή των fake news και που είναι η ελευθερία του τύπου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ψοχωρούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Συμβαστική πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 22 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απερίφθη 13 ψήφους κατά και 11 υπέρ 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 31 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 32 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 33 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 δύο τμήματα το πρώτο παρακαλώ υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα λοιπόν πρέπει να το επαναλάβουμε ηλεκτρονικά 40 πρώτο τμήμα ηλεκτρονικά αρχής ψηφοφορία πέρας Ναι, μα αλήθεια όμως δεν ήταν δυνατό να το, το διαγνώσω το αποτέλεσμα από εδώ που κάθομαι. Δεν είχατε σηκώσει χέρια. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 47 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 48 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές Έχει απορριφθεί νομίζω, αλλά το επαληθεύσουμε. Την 50 λοιπόν. Επαληθεύουμε την 50. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 16 κατά, 8 υπέρ. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη συμβαστική 8 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70, 70 υπέρ κατά. Αποχές. Απερίφθη συμβαστική 10 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ας επαληθεύσουμε 80. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 15 κατά, 9 υπέρ, απεριφθή συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 12 συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές και νομίζω ότι έχει εγκριθεί ας επαληθέψουμε όμως για να είμαστε βέβαιοι την 87 αρχίζει η ψηφοφορία 25 υπέρ, 2 κατά. Πάλι δεν σηκώσατε το χεράκι. Εγκρίνεται. 14. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά και αρχίζει. Πέρασε. 22 υπέρ. Καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Ομόφωνα δηλαδή και συγχαρητήρια θερμά στον εισηγητή μας. Να είμαστε λοιπόν Έχει μαλλιά σημαίνει γλώσσα μου, αλλά σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ εντατική και συντονισμένη δουλειά. Τελειώσαμε τις μαραθώνιες ψηφοφορίες και πάμε στο 7 στην ημερήσια Στην κανονική μας δηλαδή δουλειά, εξέταση έκθεσης πρωτοβουλίας για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλη σημασία για μας η έκθεση καθώς μάλλον έχουμε παρακαλώ παρακαλώ καθώς έχουμε λάβει την απόφαση για μια τέτοια ε, έκθεση πρωτοβουλίας βλέπουμε να τη βλέπουμε, την παρακολουθούμε να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία γιατί όλο και νέες ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατίθενται και έτσι σχετικές πάντα με την έκθεση αυτή, ενισχύεται το βάρος της. Η αγαπητή Κριστίνα Λιμπάτσικα έχει αναλάβει λοιπόν τιτάνιο έργο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, όποιο θέλει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει ήσυχα και γρήγορα για να προχωρήσουμε στη δουλειά μας κι εμείς δεν είναι προνόμιο των ολίγων η εκπαίδευση, είναι ανθρώπινο δικαίωμα, έχει στρατηγική σημασία για τις κοινωνίες μας, Το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκ τούτου δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση πλέον στην ε, εκπαίδευση από ό,τι μέχρι τώρα, παρά τις ε, ε, εθνικές αρμοδιότητες και παρά το σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες. Είναι καλό, είναι σωστό, είναι σημαντικό σε αυτό το στρατηγικό, στρατηγικό σημείο και εμείς ως Κοινοβούλιο να τοποθετηθούμε για το θέμα αυτό με τη γνωμοδότηση. Θέλω να δώσω λοιπόν το λόγο στην Κριστίνα για να μας παρουσιάσει την εκθεσή γνωμοδότησης και να περάσουμε στη συνέχεια στη συζήτηση. Κριστίνα, έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, εσάς, όλους τους συναδέλφους για την ε, συνεργασία που είχαμε, τους ε, συμβούλους πολιτικής, τη Γραμματεία, την Κομισιόν, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και θέλω να ευχαριστήσω και την βοηθό μου. Ήταν πραγματικά ανεκτήμητη η δουλειά της και θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπατε κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι ε, υπήρξαν για πρώτη φορά τόσες πολλές ανακοινώσεις της Κομισιόν για το θέμα της ε, εκπαίδευσης. Ε, χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε αυτό. Φαίνεται ότι αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα της ε, Κομισιόν η εκπαίδευση, η παιδεία. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρεθεί στην πρώτη γραμμή και να μην αντιμετωπίζει ως δευτερεύουσα σημασία στα ζητήματα της παιδείας. Και κάτι ακόμη. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ήταν να συμπυκνώσω το θέμα αυτό σε 7.000 χαρακτήρες. Μου φάνηκε σχεδόν αδύνατον αρχικός. Γι' αυτό και έχω προετοιμάσει 100 τροπολογίες που συμπληρώνουν το κείμενο και αναπτύσσουν βάσει και των τελευταίων ανακοινώσεων της Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους συναδέλφους να εξετάσουν, να διαβάσουν αυτές τις τροπολογίες και αν μπορούν να τις υποστηρίξουν. Τώρα, ως προς την ίδια την έκθεση, ε, ξεκίνησα από τρεις αφετηρίες. Πρώτον, μέχρι τούδε το σχολείο αποτελούσε το χώρο απόκτησης γνώσεων. Το ήταν το βασικό ε, η βασική πηγή ε, γνώσεων για τα παιδιά. Για μας όμως είναι σημαντικό στον χώρο εκπαίδευσης το σχολείο να μην είναι απλώς ένας χώρος απόκτησης γνώσεων αλλά ένας, ένα, ένας αξιόπιστος χώρος, ελκυστικός. Δεύτερον στόχο του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η μόρφωση των ανθρώπων και όχι μόνο η προετοιμασία των αυριανών εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες ε, των ε, ανθρώπων ως μέλη της ε, κοινωνίας. Και τρίτον, τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι και ορθώς ότι είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια για το σκοπό αυτό συνάπτονται και στρατιωτικές συμμαχίες ε, και πραγματοποιούνται και στρατιωτικές δαπάνες. Ε, με τον ίδιο τρόπο ε, θα πρότεινα εγώ να ε, θεωρηθεί και η εκπαίδευση ως τμήμα της ασφάλειας και να συναυθεί και μια αντίστοιχη μη στρατιωτική συμμαχία με αντίστοιχους σκοπούς για την έκθεση αναδεικνύουμε την ε, αποφασιστική σημασία που έχει η παιδεία και για την οικονομική ανάπτυξη. Αναφερόμαστε στις προκλήσεις των διαφόρων βαθμίδων ε, της παιδείας. Τρίτον, χωρίς δασκάλους δεν υπάρχει παιδεία. Και τέλος έχουμε κάποιες συστάσεις ε, για την Κομισιόν, για τα επιμέρους κράτη-μέλη, αλλά και για τους φορείς της εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην δημοτική εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ε, εναπόκειται ένας, ε, ανατίθεται ένας πολύ σημαντικός ρόλος, ακριβώς γιατί χαρακτηρίζει και ε, δίνει την κατεύθυνση για, τους, ε, ε, τη μετέπειτα πορεία των εκπαιδευομένων. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να αποκτώνται εκεί οι βασικότερες δεξιότητες. Δεύτερον, τα σχολεία πρέπει να αποτελέσουν κέντρα της δημιουργικής σκέψης. Και στη σημερινή εποχή, όπου πλέον αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η τεχνολογία, δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε και να θεωρήσουμε ότι η μηχανική εκπαίδευση ε, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντίθετα, η κριτική σκέψη, η δημιουργική σκέψη είναι ε, το ζητούμενο. Βεβαίως με χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για να μπορεί και να εξατομικεύεται, αν θέλετε, η εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα να αξιοποιούνται στον μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Λέμε επίσης ότι τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να υποστούν αλλαγές. Χρειάζεται και επίσης μεγαλύτερη φροντίδα για τους διδάσκοντες. Και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συμπράξεις, συνέργειες και να αξιοποιηθεί αφενός η επιθυμία των νέων ανθρώπων ε, και η τάση τους προς τις νέες τεχνολογίες με τις γνώσεις των διδασκόντων. Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Και υπάρχει ένα υπάρχει ένα δίπολο γνώση και έρευνα. Χρειάζεται όμως και ευελιξία και αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης, κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί ως έργο ακόμη. Διότι δεν αναγνωρίζονται πάντοτε ε, οι μη, τυπικές, ε, οι μη τυπικοί κύκλοι σπουδών ε, στην, στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν η γνώση και η έρευνα να αλληλοτροφοδοτούνται και να συμβαδίζουν και τέλος διδάσκοντες όλων των βαθμίδων. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα αν δεν υπάρξει ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης διδασκόντων. Οι ακαδημαϊκές γνώσεις λοιπόν βεβαίως και εξακολουθούν να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κανείς δάσκαλος ή καθηγητής. Ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητο να, ε, να μπορεί κανείς να ασκεί το λειτουργήμα αυτού. Και γι' αυτό ζητούμε να υπάρχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες στα αναλυτικά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα δίνουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε φοιτητή να απαντά «Εγώ μπορώ να γίνω δάσκαλος ή καθηγητής, έχω τα φόντα». Και ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε και τελειώνω. Αναφέρεται επίση στην έκθεσή μου ότι χρειαζόμαστε και μια θετική διαδικασία επιλογής. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σας καλώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου. Ε, βεβαίως γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, διαφορές ως προς τις των ε, Επιτροπών Πολιτισμού και Απασχόλησης. Ε, δεν αμφισβητώ καθόλου το γεγονός αυτό. Έχουμε την, ε, την γνωμοδότηση της αδέλφου Σόιντροβα, η οποία ε, συντάσσει τη δική τη γνωμοδότηση και νομίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, πράγματι, ήταν ε, εκτενής η έκθεσή σας αυτή, γι' αυτό και σας έδωσα περισσότερο χρόνο να μας την παρουσιάσετε. Και περνάμε τώρα στη συζήτηση να δώσω το λόγο στους πρώτα για δύο λεπτά το πολύ, σας παρακαλώ, η κυρία Μπόσκο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Λιμπάτσκα για την έκθεσή της. Την έχει διατυπώσει πολύ σωστά. Είναι ένα πολύ εμπεριστατωμένο έγγραφο, εξαιρετικό. Δεν υπάρχουν και πολλά που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Συμφωνώ με τη δομή με την αρχιτεκτονική του κειμένου τονίζει όλα τα επίπεδα, όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Χαίρομαι, διότι αναφέρεται και στην ε, προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι ένα πολύ επαγγελματικό έγγραφο, το οποίο προέκυψε μετά από συναντήσεις με πολλούς εκπροσώπους του κλάδου. Ε, είναι μια πολύ ολοκληρωμένη δουλειά. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το γεγονός ότι πράγματι δεν υπάρχει μια ομοιόμορφη λύση που μπορούμε να εφαρμόσουμε παντού, μια μαγική συνταγή που θα λειτουργήσει αμέσως σε κάθε κράτος μέλος και σε κάθε κατάσταση. Το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές, να τις διαδίδουμε και η επένδυση στην εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική. Όσες χώρες επενδύουν στην εκπαίδευση και στον εξυγχρονισμό αυτής, σημειώνουν πρόοδο, αναπτύσσεται η νεολαία τους, αναπτύσσεται η οικονομία. Άλλωστε, η εκπαίδευση των διανοουμένων θα οδηγήσει σε μια κοινωνία στην οποία οι πολίτες θα έχουν δεξιότητες αγωγής του πολίτη και θα έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση, θα είναι μια κοινωνία πολύ πιο ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος. Ως προς τα σχολεία, η συνεργασία με τους γονείς είναι εξαιρετικά σημαντική και με την τοπική και περιφερειακή κοινότητα και τις οργανώσεις των νέων. Θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνεργασία. με τις 100 τροπολογίες. Με πολλές από αυτές συμφωνώ και θα τις υποστηρίξω. Αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει είναι το εξής. Μία διατύπωση που θα λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, των φοιτητών που ε, θα γίνουν καθηγητές και ε, να ε, ε, ε, συνεχίζουμε την εκπαίδευση των μητέρων και των οικογενειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και περνάμε στον κύριο Σερνατζότο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση δεν μπορούμε να αφήσουμε τα κράτη μόνα τους, ούτε την κατάσταση να συνεχίζει να ε, έχει έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μία και καινία φωνή για την εκπαίδευση, για την προσχολική ηλικία. Πιστεύω ότι πραγματικά τονίσατε και αναδείξατε τα σωστά ζητήματα, τα πιο επίκαιρα. Με ενδιαφέρει η τροπολογία 57 που αναφέρεται στο ρόλο κλειδί των γονέων. Δηλαδή οι γονείς κάνουν εκπαιδευτικές επιλογές και αυτό είναι σημαντικό και θα υποβάλουμε τροπολογίες για τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν. Η οικογένεια είναι μια δομή, μια μικρή κοινότητα, ένας πυρήνας στη ε, κοινωνία. Εάν δεν ξεκινήσουμε από την κοινωνία θα πάμε σε ένα κράτος το οποίο θα είναι ανώτερο μεν, θα υπερισχύει στην ιεραρχία, αλλά δεν θα έχει κοινότητες από κάτω του να στηριχθεί. δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε από τις οικονομικές δυνατότητες. Δηλαδή, μια οικογένεια με ε, περιορισμένα οικονομικά μέσα δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε λιγότερη εκπαίδευση λόγω αυτού. Η Ευρώπη που μας αρέσει γιατί η, σημερινή Ευρώπη δεν μας αρέσει καθόλου έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη που μας αρέσει όλα αυτά θα τα περιλαμβάνει. Μιλούμε για το δικαίωμα των νέων, των παιδιών, των εφήβων, των ενηλίκων, των νέων ενηλίκων να επιτύχουν αυτό το στόχο, να έχουν πρόσβαση σε μια όσο δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Επομένως η έκθεση σωστά λέει ότι είναι σημαντικό ε, μέσα από την εκπαίδευση να δημιουργείται το άτομο, να δημιουργείται ο πολίτης, ένας πολίτης. Και μετά θα πρέπει κανείς να έχει την κατάλληλη εκπαιδευτική διαδρομή για να μπορεί να βρει μια θέση απασχόλησης. Αλλά δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση μόνο ως προετοιμασία για κάποια απασχόληση. Η εκπαίδευση είναι και προετοιμασία για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του πολίτη. Δεν θα αλλάξουμε δομικά στοιχεία αυτής της έκθεσης, αλλά θα υποβάλουμε τροπολογίες σχετικές. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια παρακαλώ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Κριστίνα Λιμπάτσκα γιατί έχουμε πολύ στενές σχέσεις. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτή, θέλησε να επικοινωνήσει ιδιαίτερος μαζί μας, να δεχθεί τις προτάσεις μας. Ήταν πολύ εύκολο πραγματικά να συνεργαστούμε. Εμείς συμφωνούμε με πολλά από τα περιεχόμενα της έκθεσης, έχουμε πολλά κοινά. Η εκπαίδευση είναι κάτι το θεμελιώδες και παρόλο που είναι αρμοδιότητα των κρατών μαελών, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να μπορεί να ε, βοηθήσει και να μπορεί να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το πάρει στα σοβαρά. Μιλούμε για ποιοτική εκπαίδευση που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη μιας ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης με Ευρωπαίους πολίτες ενεργητικούς δραστήριους που συμμετέχουν ενεργητικά στο ε, ε, ευρωπαϊκό οικοδόμημα για να έχουμε τις κατάλληλες κοινωνικές δομές και να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σημείο εστίασης θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μας οι καθηγητές, η κατάρτισή τους, η απόκτηση δεξιοτήτων για να μπορέσουν να βγάλουν το καλύτερο που έχει ο κάθε μαθητής μέσα του, να μπορέσουν να το βγάλουν προς τα έξω. Και το ταλέντο είναι σημαντικό. Επομένως, για να έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο και ποιοτικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ατομικές διαφορές. Δεν έχουν όλοι οι μαθητές τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ικανότητες για μάθηση, το ίδιο ταλέντο και τις ίδιες ακριβώς ε, ε, ιδιότητες. Υπάρχει πολυμορφία και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη φαιά ουσία των μαθητών μας, οι οποίοι καλούνται να υπάρχουν σε ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντική η διδασκαλία της κριτικής σκέψης στο σχολείο. Με αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί Μιλούμε ε, για την εποχή των fake news, των ψευδών ειδήσεων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορεί ο κόσμος να έχει κριτική σκέψη και να τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα καταλάβουν και να τα αντιληφθούν οι μαθητές αν έχουν ήδη διδαχθεί εργαλεία κριτικής σκέψης. Βεβαίως ε, πρέπει να δώσουμε έμφαση για τις απαραίτητες, στις ικανότητες και διορθώσεις ε, της εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκρίνεται και στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κόρτσο Μαλτέζα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κατερίνα, την Κριστίνα Λιμπάτσικα, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά, ψηλού επίπεδου. Είναι όλο αυτό το θέμα για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης που έχει εκφυλιστεί τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα η παράγραφος εκείνος, εκείνο που αναφέρεται στην ε, κατάρτιση πολιτών και όχι εργαζομένων ή εργατών από την εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι κάτι το οποίο νομίζω εκφράζεται σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά συντάγματα. Τα τελευταία χρόνια ο εξυγχρονισμός έγινε αντιληπτός ως μια εκλαϊκευμένη μορφή χειραγώγησης του κλασικού δημόσιου σχολείου. Έτσι ώστε αυτό αντί να παράγει, αντί να μορφώνει ε, πολίτες με κριτικό πνεύμα, να κατασκευάζει μυρμηγκάκια που θα δουλέψουν, θα βγουν στην αγορά της εργασίας. Ε, νομίζω ότι με αυτό το πνεύμα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ε, προσέγγιση της ε, συναδέλφου Λιβάτσικα. Πρέπει να εξυγχρονιστεί βεβαίως το σχολείο, γιατί κινδυνεύει να ξεπεραστεί από τη νέα κοινωνία της τεχνολογίας, εάν δεν εξυγχρονιστεί. Και ο δρόμος είναι αυτός τον οποίο υποδεικνύει η συνάδελφος. Εμείς μόνο κάποιες τροπολογίες που ενισχύουν τις πτυχές της ενσωμάτωσης των προσφύγων, παραδείγματι, και, του, και την έμφαση στο κριτικό και δημιουργικό πνεύμα έχουμε να εισαγάγουμε. Βεβαίως, πολύ σημαντικό, εάν θέλουμε ακριβώς να μορφώσουμε πολίτες με κριτικό πνεύμα και με συνείδηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Μπίλτ, Μπίλντε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είχε φιλοδοξίες καινοτομία, αλλά το μόνο που κάνει είναι αναμασά τα στερεότυπα που κάνουν την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πέφτει συνεχώς στην κατάταξη πίζα και οι χώρες που έχουν τις ε, μεγαλύτερες επιδόσεις ε, στο σύστημα PISA δεν είναι ε, αυτές που βάζουν την παπαγαλία και το να μαθαίνουν πράγματα απ' έξω. Κίνα και άλλες χώρες έχουν υψηλότερες επιδόσεις, παρόλο που δίνουν λιγότερο ποσοστό του ΑΕΠ στην παιδεία. Η Φιλανδία έχει πέσει 10 θέσεις στα μαθηματικά στην κατάταξη PISA και 11 θέσεις στις επιστήμες, από το 11 μέχρι το 12, το 2011 μέχρι 12. Οι Φιλανδοί εμπειρογνώμονες εν μέρη αποδίδουν αυτή την οπισθοχώρηση στην υποδοχή των μεταναστών και στις νέες τεχνολογίες που κάνουν τα νέα αγόρια κυρίως να διαβάζουν πολύ λιγότερο και να κάνουν πολύ λιγότερη ανάγνωση. Στη Γαλλία πριν από 25 χρόνια είχαμε προσπαθήσει να σταματήσουμε να μαθαίνουμε ε, στα παιδιά ε, την προπαίδεια απ' έξω και μέχρι, μετά από τρία-τέσσερα χρόνια καταλάβαμε ότι ήταν τεράστιο λάθος, γιατί αφού δεν ήξεραν υπό την προπαίδεια δεν μπορούσαν να κάνουν και υπολογισμούς με το μυαλό τους ε, τα παιδιά και τελικά ε, γυρίσαμε στην αρχή και δεν προλάβαμε αυτές τις γενιές, δύο-τρεις τάξεις που έγιναν ενήλικες και δεν είχαν διδαχθεί την προπαίδεια, δεν την είχαν μάθει απ' έξω. Δεν θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον πύχη, υποδεχόμενοι παιδιά με πολύ χαμηλό επίπεδο στο, όπως οι μετανάστες. Σε κάθε περίπτωση, σε όλα αυτά τα ζητήματα προβλέπεται όλα αυτά τα οποία δεν πρέπει κανείς να κάνει και είναι λάθος. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες παρόλο που δεν θα τύχουν και ευρεία στήριξη από την πλειοψηφία ω συνήθω Αλλά έχουμε την υποχρέωση να το πράξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πριν προχωρήσουμε στις επόμενες παρεμβάσεις. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω μια ομάδα επισκεπτών στην Επιτροπή μας. 13 επισκέπτες από το Απρούτσο της Ιταλίας, από διάφορες ε, κοινότητες και χωριά του Απρούτσο. Προσκεκλημένοι του Μάσιμο Παολούτσι, του Ιταλού. Συναδέλφου, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και ελπίζω να ακούτε κάτι το ενδιαφέρον κάτι που θα μπορέσετε να μεταφέρετε και στην Ιταλία. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ακούμε τους λοιπούς συναδέλφους. Ο κύριος Σβεά, δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λιμπάτσκα για την πολύ καλή της δουλειά, για την έκθεση αυτή. Και τους άλλους κοιόδης εισηγητές και την κυρία Πόσκο, εισηγητρία από την ομάδα μου. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει διάφορα έγγραφα για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την ανανεωμένη ατζέντα για την επένδυση στους νέους της Ευρώπης, για την ανώτερη εκπαίδευση, την τριτοβάθμια. Στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης αναφέρεται η εκπαίδευση επίσης. Έχει σημαντικό χώρο να καταλάβει με θεωρείται σου και είναι ευρέως γνωστό ότι η εκπαίδευση συμβάλλει η ποιοτική στην ανάπτυξη, στη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Οι νέε πολιτικέ ε, στον τομέα τη εκπαίδευση είχαν σημειώσει αρκετή επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Ο στόχο είναι το 40% των νέων να έχουν ε, αποκτήσει, να έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2020 και είμαστε κοντά σε αυτό το στόχο. Ε, όμως αυτό που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αναντιστοιχία μεταξύ ε, δεξιοτήτων που έχουν οι μαθητές οι φοιτητές και αυτό που ζητείτε. Δηλαδή, πολλοί αποφυτούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με πολύ φτωχές δεξιότητες και με δεξιότητες που δεν μπορούν να ε, εφαρμόσουν διατομεακά, δηλαδή, για παράδειγμα, εργαλεία επίλυσης προβλημάτων ευρύτερων και αυτό δεν συμβάλλει στο κλίμα του επιχειρήν και στην καινοτομία στην στην οικονομία. Χρειάζεται περαιτέρω εξυγχρονισμός από την αρχική προσχολική εκπαίδευση και κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα είναι τα πιο ελκυστικά μέρη στο σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο. Έχουμε τους παραδοσιακούς χώρους μάθησης που συμπληρώνονται από πολλές άλλες πηγές πληροφόρησης με τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως πολύ σωστά τονίζει η συγγήτρια. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της Μπολόνιας, να ενοποιήσουμε τον χώρο τρίτος βάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα σχολεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σοϊντρόβα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω πάνω απ' όλα να εκφράσω την ε, τη σημασία που έχει εκθέσει συναδέλφου. Είναι πάρα πολύ καλή και θα πρέπει να την μελετήσει διεξοδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι έχω πιο επικριτικό βλέμμα από τη συνάδελφο προ τη συμπεριφορά, τη στάση τη Επιτροπή στο θέμα αυτό. Άλλωστε και την εκφράζω και θέλω να υπογραμμίσω και εγώ τη σημασία του σχολείου, τη σημασία του διδακτικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, τη ε, κατάρτιση στο σημείο 13 έω 16. Εκεί όπου μιλούμε για τη σχολική εκπαίδευση, πρέπει να τονιστεί η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση και της τεχνικής κατάρτισης. Τα new skills επίσης έχουν μεγάλη σημασία, όπως το αναφέρει η συνάδελφος. Αλλά δεν είναι σαφές ε, το εάν είναι ικανοποιημένη συνάδελφος από τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτελεί το σχετικό έργο, εάν δηλαδή κάνει αυτό που όφιλε. Έτσι λοιπόν το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες, new skills, θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού συστήματος ε, και στον εξυγχρονισμό του ενώ εδώ βλέπουμε μια νέα εκδοχή της διαδικασίας της Ορβόνης, αναγνώριση δηλαδή των πτυχίων και απολυτηρίων, κάτι το οποίο σχετίζεται και με τη διαδικασία της Μπολόνια. Και άρα το πρώτο και κύριο είναι να εξελιχθεί περαιτέρω, να αναπτυχθεί περαιτέρω η διαδικασία της Πολώνια, γιατί δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη, δεν δίνει τα ίδια αποτελέσματα, δεν, δίνει, δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τι εργαλεία πρέπει να έχουμε στη θέση μας όσοι δεν έχουν το, τα εργαλεία της ε, Πολώνια Ευχαριστώ τη συνάδελφο. Πρέπει να προβάλλουμε και να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόκληση αυτή να κάνει τη δουλειά της όπως οφείλει. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μοργάνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την Κριστίνα για το έγγραφο που μας έχει υποβάλει. Δεν πρόκειται για ευχαριστίε ε, για λόγου απεφροσύνης. Είναι ουσιαστικέ ευχαριστίες μου, γιατί νομίζω ότι εδώ ερχόμαστε να δώσουμε απαντήσει σε μελλοντικέ προκλήσεις. Ε, και γιατί λαμβάνω το λόγο, γιατί η υποχρέωση σε 7.000 χαρακτήρες, τυπογραφικούς χαρακτήρες να περιορίσουμε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα, θέμα τεράστιο κόπο και μόχθο και ήδη το γεγονό ότι καταρτίστηκε αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική από την εισηγήτρια. Εγώ προσωπικώς θα εμβαθύνω όσο μπορώ στο θέμα. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμο, όπως άλλωστε έχουμε ήδη συζητήσει και υπενθύμησε και η Πρόεδρος, να υπογραμμίσουμε, να επιστήσουμε την προσοχή σε σχέση με το θέμα με τη σημασία του σχολείου και της ε, σχολικής μόρφωσης και πέραν και των ε, αρμοδιοτήτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε εις βάθος τα θέματα που θα προκύψουν και σε σχέση με τις συστάσεις του κειμένου της Κριστίνα. Η προσπάθεια για μία προσέγγιση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ε, ανάπτυξης ενός κοινού δυναμικού των εκπαιδευτικών και βέβαια το θέμα τη προετοιμασία για την αγορά εργασία. Αυτό όμω τι σημαίνει, τι σημαίνει, ποια είναι η αγορά εργασία στην οποία αναφερόμαστε η τωρινή, η μελλοντική που δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει λάβει. Τι σημαίνει αυτή η εκπαίδευση. Πολλέ είναι οι πτυχέ που ήδη υπενθύμησε η Κριστίνα, οι ανθρωπιστικέ πτυχέ που θα πρέπει να τονιστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, σε ένα σημείο που δεν είμαι βέβαιος αν έχω αντιληφθεί σωστά το, τη σύσταση, ε, ίσως να είναι θέμα στη μετάφραση βέβαια. Τι σημαίνει πρώτη παιδική ηλικία ή βρεφική ηλικία, ενώ από τα 0 μέχρι τα 7 χρόνια, από τα 2 μέχρι τα 7, 4, 5. Ε, ας το ορίσουμε αυτό, δεν είναι πολύ σαφές. Γιατί ανάλογα βέβαια εξαρτάται και τι είδος ε, σχολικού πλαισίου ε, μας ενδιαφέρει. Αυτά λοιπόν, ε, λίγο πολύ, αυτές θα είναι και οι τροπολογίες μου προκειμένου να ενισχύσω το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ και πριν του δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια. Θα παρακαλέσω την Επιτροπή, ε, τον κύριο Τόιτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Θα ήθελα να επανέλθω στην αρχή της συζήτησης όταν υπόθηκε ότι πράγματι η Κομισιόν ε, έχει επιδείξει μια πολύ μεγάλη φιλοδοξία στον τομέα της εκπαίδευσης της παιδείας. Υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία, νέες ανακοινώσεις και ε, έχουμε πλέον σαφή τη θέση ότι παρά τις εθνικές αρμοδιότητες πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ε, ε, παιδείας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται για την παιδεία ή για την εκπαίδευση επειδή δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς επειδή έχει ως στόχο της την κοινωνική συνοχή που έχει και μια κοινωνική και πολιτιστική διάσταση και εκπαιδευτική βεβαίως ε, έχει κάθε λόγο να ε, δραστηριοποιείται στον ε, τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της ενίσχυσης ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γι' αυτό και ευχαριστούμε για αυτή την έκθεση. Υπάρχουν εξελίξεις και στον τομέα του, του Εράσμους, βεβαίως θα συζητηθούν. Μπορούμε να κάνουμε φυσικά περισσότερα πράγματα, έχετε δίκιο σε αυτό να απαντήσω ε, για τα, στα σχόλια. Προσχολική ε, αγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι υψηλής ποιότητας η, η προσχολική αγωγή. Ε, όταν μιλούμε για ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, δεν είναι μόνο ένας χώρος ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από κινητικότητα, αλλά και από υψηλή ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στην υψηλής ποιότητας προσχολική αγωγή αφενός και την αναγνώριση αφετέρου του πολύ σημαντικού ρόλου που παίζουν οι οικογένειες. Οι οικογένειες σε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις σήμερα διαδραματίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλλον διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υψηλού επίπεδου υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και των παιδών, δεν, ε, παιδιών. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίθεση μεταξύ των δύο. Ε, εκπαίδευση διδασκόντων, καθηγητών, δασκάλων. Φυσικά μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα ε, τον ε, Ιανουάριο μάλιστα ε, υποβάλαμε και μια δέσμη προτάσεων, ε, συστάσεων μάλλον για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και τέλος για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Τι είναι ο, χώρος αυτός. Δουλέψαμε πολύ, αλλά μια και αναφέρθηκε και η Μπολόνια, πρέπει να σας πούμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώθηκε. Ε, παρά την πολύχρονη ε, συνεργασία και την Πολόνια υπάρχει ακόμα, υπάρχουν ακόμα πολύ σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων, πτυχίων. Ε, γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα, τα εμπόδια, να καταργηθούν φραγμοί που υπάρχουν ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην κινητικότητα των νέων ανθρώπων στην έβρεση εργασίας, στην έβρεση ε, δυνατοτήτων και ευκαιριών ε, εκπαίδευση. Γι' αυτό και χαιρόμαστε πολύ για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Κριστίνα, έχει το λόγο. Προσπάθησε παρακαλώ, αν γίνεται, σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρία σημεία. Σε κάθε βαθμίδα υπάρχουν, υπάρχει ένα τρίγωνο. Μαθητές, διδάσκοντες και γονείς. Και πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των ε, τριών πλευρών. Θέλω να καθησυχάσω όλους όσοι είπαν ότι δεν λαμβάνω υπόψη μου τους γονείς. Αντίθετα, βεβαίως η εκπαίδευση είναι εθνική αρμοδιότητα. Όμως, κοιτάξτε το πρόγραμμα Erasmus+. Πόσο εξαιρετικά αποτελέσματα έχει αποφέρει αυτή η ανταλλαγή φοιτητών Μιλούμε για εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, για την ευρωπαϊκή και δημιουργική σκέψη, μα απαραίτητο στοιχείο για κάτι τέτοιο είναι η κινητικότητα εκπαιδευομένων και διδασκόντων, αλλά και η κατάρτιση προδιαγραφών ποιότητας για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Και τρίτον, πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι μαθητές και φοιτητές ε, παρουσιάζουν πολλές διαφορές μεταξύ τους. Πράγματι, Γι' αυτό και αναφέρουμε στην έκθεση ότι χρειάζεται εξατομίκευση των, ε, της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και γι' αυτό και υπησέρχομαι στην, στην έκθεση αυτή ε, σε μια σειρά από θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο και των ανακοινώσεων. Θα, θα, τα εντάξω αυτά τα θέματα και μέσω των τροπολογιών βεβαίω, γιατί δεν είχα την ευκαιρία στο σώμα του κειμένου να τα ε, συμπεριλάβω όλα. Θέλω για να πω και κάτι τελευταίο. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, για τις, ε, ε, για τις απόψεις που ακούστηκαν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα να ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Κομφούκιου, της Άπο Ανατολής, όπου που βεβαίως είχε και έκφραση και στην αρχαιοελληνική σκέψη. Τι, τι θέλω να πω. Πρέπει ταυτόχρονα με τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους να διατηρήσουμε τον, τον πυρήνα ε, της ε, παραδοσιακής μας σκέψης ότι στο κέντρο της εκπαίδευσης είναι η σχέση του διδάσκοντα με τον μαθητή του. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 28 Φεβρουαρίου ψηφοφορία θα γίνει 25 Απριλίου και κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην πολύ σημαντική αυτή έκθεση που έχετε αναλάβει. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη έκθεση που είναι η υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Νεολαία η κυρία Γκάρδια Ζαβάλ είναι η Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στην Άιντα και μετά θα προχωρήσουμε στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω την έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ ως προς την νεολαία. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στο μέλλον είναι να καταφέρουμε ε, η νεολαία να γίνει εγκάρσια πολιτική και να είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε τώρα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής στο μέλλον. Μιλούμε για τις βασικές γραμμές εργασίας, όπως για παράδειγμα η άμυνα ή το περιβάλλον ή η έρευνα. Όταν όμως μιλούμε για τους νέους, δεν μιλούμε για τους νέους ως γενική και εγκάρσια πολιτική, αλλά ε, επιλεκτικά κατακαιρματισμένα προγράμματα όπως είναι το Εράσμος ή η εγγύηση για τους νέους και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι συμπτώματα που δείχνουν ότι δεν έχουμε πραγματικά αφομοιώσει ότι η πολιτική για την νεολαία πρέπει να είναι εγκάρσια, δηλαδή να αφορά όλες τις υπόλοιπες πολιτικές και να τις διατρέχει. Σιγά σιγά φαίνεται αυτό στις πολιτικές ομιλίες, αλλά θα πρέπει ε, τις πολιτικές ομιλίες να τις μεταφράσουμε σε συγκεκριμένες στρατηγικές πράξεις τα επόμενα χρόνια. Και με αυτό το στόχο λοιπόν έχω χωρίσει την έκθεσή μου σε πέντε κεφάλαια και έχω προσπαθήσει να αναλύσω πώς λειτουργήσε η στρατηγική για την νεολαία, προτείνοντας συνάμα δράσεις για τη βελτίωση της στρατηγικής στο μέλλον. Το καλύτερο με τη στρατηγική αυτή ήταν ότι ήταν μια καλή βάση για επικοδομητική συνεργασία. Θέσαμε κοινούς στόχους, κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, χρηματοδότηση και ε, ε, διαρθρωμένο δομικό διάλογο για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των νέων. Η στόχη όμως ήταν εξαιρετικά γενική και δεν έχουμε αρκετούς δείκτες και κυρίως κοινούς δείκτες για να μπορούμε να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο αυτής της στρατηγικής. Μεταξύ των θεμάτων που αναδεικνύω είναι εισαγωγικά καταρχάς να πω τα εξής η φωνή και η συμμετοχή των νέων. Εάν θέλουμε μια στρατηγική πραγματικά να λειτουργεί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νεολαία, οι ενώσεις, οι σύλλογοι, όλες οι οργανώσεις των νέων να είναι μέτοχοι στην αξιολόγηση, στην εκπόνηση και στην εφαρμογή των πολιτικών ε, των νέων μέσα από τα διάφορα εργαλεία είναι υποχρέωση της δημόσιας εξουσίας να δώσει τη δυνατότητα και να ενθαρρύνει την νεολαία να συμμετάσχει περισσότερο και να νιώσει πιο εμπλεγμένη, πιο ε, δρόν παράγοντας, αν θέλετε, στα της κοινωνίας. Και ένα από τα βασικά είναι η απασχόληση βέβαια. Ξέρουμε ότι τα ποσοστά απασχόλησης των νέων έχουν βελτιωθεί όμως η ενεργεία των νέων κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και πρόκειται για απασχόληση αβέβαια, ε, πολύ περισσότερο αβέβαια από ότι σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Είναι επαναληπτικό, αλλά δεν μπορούμε να μην το επαναλάβουμε ξανά και ξανά, ότι δίνουμε έμφαση στην ποιοτική εργασία των νέων, στα εργασιακά τους δικαιώματα, στα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα, γιατί η σημερινή απασχόληση έχει να κάνει, συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία όμως δεν τα έχει η νεολαία και τις τα στερούμε. Τρίτο θέμα με, που σχετίζεται με την νεολαία είναι η εκπαίδευση. Βεβαίως μόλις τώρα είχαμε μια συζήτηση πολύ μακροσκελή για τα της εκπαίδευσης και δεν πρόκειται να σας δώσω λεπτομέρειες για το τι υπάρχει στην έκθεση σε σχέση με την εκπαίδευση. Είναι από τους βασικούς πυλώνες η εκπαίδευση για την πολιτική για την νεολαία. Απασχόληση είναι ο ένας πυλώνας, εκπαίδευση ο άλλος για την στρατηγική για την νεολαία. Τα έχω τονίσει αρκετά αυτά και θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον να ανοίξουμε και νέα πεδία εργασία στην έκθεση, γιατί δεν είναι μόνο η απασχόληση και η εκπαίδευση πυλώνες της πολιτικής για την νεολαία. Η πολιτική για την νεολαία επηρεάζεται και από άλλες περιοχές και από άλλους τομείς επίσης. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει εγγύηση για τα παιδιά. Ε, όχι μόνο για τους νέους, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ευκαιρίες στο μέλλον. Αγωγή του πολίτη, σεβασμός, ανεκτικότητα, ανεξιθρησκεία, ανοχή, αξίες που θέλουμε να διαδώσουμε στην νεολαία και να τις σφυριλατήσουμε. Και υπάρχει και το θέμα της παρενόχλησης και της κυβερνοπαρενόχλησης του μπούλιν αλλά και ε, του ε, ιντερνετικού μπούλιν και το θέμα της ψυχικής υγείας, τα επίπεδα στρες και άγχους των νέων ε, αυξάνονται, πρέπει να τους βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Και τέλος υπάρχει και το θέμα της κουλτούρας και του πολιτισμού γιατί αυτό είναι το, ο μεγαλύτερος φραγμός, το μεγαλύτερος προμαχώνας για την υπεράσπιση έναντι της μυσαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και το καθεξής. Και τέλος χρηματοδότηση. Πώς θα χρηματοδοτηθούν και ποια θα χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση τα προγράμματα που έχουν ταυτιστεί με την πολιτική νεολαίας δεν χρειάζεται να τα υπερασπιστούμε, γιατί τα αποτελέσματά τους μιλούν από μόνα τους, δείχνουν εύγλωτα από μόνα τους την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. Άρα είναι δίκαιο να ζητήσουμε ενίσχυση της χρηματοδότησης και για την Ευρώπη που δημιουργεί και για την Ευρώπη για τους πολίτες και τους νέους και για την εγγύηση για τους νέους και για το πρόγραμμα Εράσμους. Όλα αυτά τα προγράμματα δεν χρειάζεται να αποδείξουμε γιατί απαιτούμε αύξηση της χρηματοδότησής τους. Επομένως, αυτό είναι μια σύντομη περίληψη με το περιορισμό της έκτασης ε, που είχαμε ε, της έκτασης της έκθεσης που μας είχε επιβληθεί προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και ευχαρίστω να δεχθούμε τροπολογίες για να διευρύνουμε και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο ε, τη διατύπωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. ηγητές. Ο κύριος Μάλινοφ τώρα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τη συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Είναι ένα πολύ καλό υπόβαθρο για τη μελλοντική μας εργασία. Χαίρομαι με τον τρόπο που οργανώνετε τα προβλήματα. Η δομή της έκθεσής σας είναι πάντοτε ο καλύτερος ε, τρόπος ε, ε, να υπάρχουν πέντε κεφάλαια και έτσι στο επόμενο στάδιο μπορούμε να δουλέψουμε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να υπενθυμίσω ότι αυτή είναι μια πρώτη αξιολόγηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που ξεκίνησε, που λασταρίστηκε. Δυσκολευθήκαμε να αξιολογήσουμε αυτή την στρατηγική γιατί δεν περιλαμβάνει πολύ σαφείς δείκτες και είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό ως θέση, αλλά και ως μελλοντικό πλαίσιο αναφοράς. Δηλαδή, χρειαζόμαστε περισσότερους δείκτες, περισσότερα απτά στοιχεία για να μετρήσουμε την επιτυχία της στρατηγικής. Πολλοί ήταν πολύ επιφυλακτικοί όταν ξεκίνησε αυτή η στρατηγική και εγκαινιάστηκε. Γιατί όλα αυτά ε, τα στοιχεία όλα αυτά τα κονδύλια μπορούν να διοχετευθούν σε διαφορετικές πολιτικές. Εκπαίδευση, άθληση, υγεία. Χρειαζόμαστε πολιτική για την νεολαία, στρατηγική για την νεολαία. Έθεταν το ερώτημα η επιφυλακτική και δείξαμε ότι είναι σημαντικό ε, γιατί και πράγματι χρειαζόμαστε τέτοια στρατηγική γιατί δόθηκε δημόσιος χώρος στους συμμετέχοντες, στις οργανώσεις των νέων. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για να τα αξιολογήσουμε. Όχι μόνο για να αξιολογήσουμε τα πρακτικά αποτέλεσματα που δυστυχώ δεν τα έχουμε ακόμα και γι' αυτό δεν τα έχουμε αξιολογήσει, αλλά είναι σημαντικό γιατί οι συμμετέχοντε το βρήκαν ιδιαίτερα χρήσιμο. Και αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη στρατηγική, Πόσο οι συμμετέχοντες είπαν ότι του βοήθησε. Ε, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τους νέους είναι ένα πράγμα και οι διατομεακές πρωτοβουλίες είναι κάτι το διαφορετικό και είναι δύσκολο να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση και να ε, κάνω και ένα ερώτημα. Γι' αυτό σας παρακαλώ μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Ε, η παιδική εγγύηση, η εγγύηση για τα παιδιά, αναρωτιέμαι, αξίζει να θεωρηθεί, να αναφέρεται εδώ. Εγώ έχω αντίρρηση επί της αρχής. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι στη στρατηγική για την νεολαία, παρόλο που είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στα σπάραγανα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα η Επιτροπή να μας πει τα επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης μιας τέτοιας αναφοράς σε αυτό το κείμενο. Και ελπίζω ότι θα προσφέρω μια λύση στο εξή πρόβλημα. Πολλοί νέοι δεν θα δέχονταν την ιδέα της ε, ιδιότητας της, ε, του πολίτη, της ε, το, το θεωρούν ως βάρος, δηλαδή να είναι κάτι, ένας πολίτης ενεργητικός, δραστήριος πολίτης, το θεωρούν ως βάρος και όχι ως μια ιδιότητα ποιοτική. Πώς θα πείσουμε τους νέους ότι όλα αυτά σχετίζονται με τις ελευθερίες, με τα δικαιώματά τους δεν είναι καθόλου προφανές ότι οι νέοι θα είναι ενθουσιώδεις με το να αποκτήσουν ακόμα πιο ενεργά την ιδιότητα του πολίτη και δεν θα την αντιλαμβάνονται ως βάρος. Ευχαριστώ. πράγματι, πρέπει να υπάρχει μια ισότητα προς τις υποχρεώσεις του και το δίκαιο πάντοτε. Ε, η κυρία Μίχελς, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον την συγγήτρια ε, για την ε, έκθεσή της, ιδίως όσον αφορά την συγκρισιμότητα των εμπειριών και την μέτρηση των αποτελεσμάτων ε, της υλοποίησης της στρατηγικής στα κράτη-μέλη. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε διοργανώσει και μια ακρόαση και εκεί καταγράφηκε και ε, το πρόβλημα σχετικά με την ε, μη δεσμευτικότητα των στόχων. Επίσης, αναδείχθηκε το θέμα των ε, περικοπών, των δαπανών στην στρατηγική για την νεολαία στα κράτη-μέλη και η διαρκής προσπάθεια ανάπτυξης των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική για την παιδεία και την νεολαία. Επίσης, χρειάζονται προϋποθέσεις, χρειάζεται πλαισίωση για να μπορεί κανείς να συμμετέχει στο δημοκρατικό πολίτευμα και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ε, ε, ενίσχυση ιδίως των ψηφιακών δυνατοτήτων συμμετοχής. Τέταρτον, ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες των μειονοτήτων, αλλά και η αυξανόμενη ανάγκη σχετικά με την ένταξη μεταναστών και προσφύγων. Και τέλος ε, χαιρετίζω την ε, ε, διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που υπερβαίνει και τα στενά όρια αυτής της στρατηγικής για την νεολαία. Και από αυτή την άποψη χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε με την συγγήτρια. Θα συμμετάσχουμε και θα υποβάλουμε και εμείς, ε, θα συμβάλλουμε και εμείς στη συζήτηση. Η κυρία Μπίλτ, αν θέλετε, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι λύσεις που προτείνετε είναι κάπως ε, προβληματικές, θα έλεγα οι νέοι για πρώτη φορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Οι λύσεις σας είναι γελίες. Δεν είναι το πρόβλημα να βρουν μια πρώτη απασχόληση ή μια πρώτη εθελοντική συμμετοχή όπως είναι στο Ευρωπαϊκό Σώμα Ελληνικής. Δεν πρόκειται να μάθουν και τίποτα χρήσιμο από αυτά τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά εργασίας. Το πρόβλημα είναι πώς θα βγουν από το φαύλο κύκλο των ε, πήγαινε έλα μεταξύ μιας ε, μικροδουλειάς και του Ταμείου ανεργία και του να μένουν με τους γονεί του γιατί δεν μπορούν να ε, ε, κάνουν κάτι άλλο. Σήμερα στη Γαλλία στα 30 τους μπορούν να αποκτήσουν μια σταθερή δουλειά. Δέκα χρόνια και ε, σέρνονται από τις εθελοντικές απασχολήσεις και τις και τα συμβόλαια μερικής απασχόλησης ή ε, προσωρινής εργασίας. Μέχρι τα 40 δεν μπορούν να φτιάξουν οικογένεια. Ε, είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα. Όταν εγώ ήμουν νέα δινόταν έμφαση στη μαθητεία, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο επιτρέπει επίσης και στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτισμού μας να ε, φανούν και οι διαφορές των κρατών μελών, οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, της κάθε εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους. Να μπορέσουν οι νέοι να ακολουθήσουν το δρόμο που έχουν ανοίξει οι γονείς και οι παππούδες τους και να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο και για τα δικά τους παιδιά όταν και αν θα τα αποκτήσουν. Σας ε, ε, εκπλήσει το γεγονός των χαμηλών ποσοστών γεννητικότητας ε, στην Ευρώπη και αυτό είναι και το φανταστικό το τρομερό πρόσχημα για να ανοίξετε διάπλατα τις πόρτες της μετανάστευσης. Δίνετε ψίχουλα στους νέους και η ελπίδα που τους δίνετε το μόνο που κάνει να τους απογοητεύει γιατί διαψεύδεται ικτρά. Ευχαριστώ. Κοιτάω στην αίθουσα Κομισιόν. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για τις απόψεις τους. Επιτρέψτε μου καταρχάς να καλωσορίσω το γεγονός, να εκφράσω την ικανοποίησή μου το γεγονός, για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ε, έχει αυτή τη συζήτηση και κάνει μια ολόκληρη συνεδρία γιατί το απασχολεί το μέλλον των νέων και συμφωνούμε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ επίκαιρο αυτό γιατί τώρα σκεφτόμαστε να ανανεώσουμε την ε, στρατηγική για τους νέους, άρα σε αυτό το πλαίσιο ε, είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση από τη στιγμή που γίνεται και η διαπραγματεύση για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι προοπτικές των νέων είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Συμφωνούμε. Τα θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά η συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες και στη λήψη των αποφάσεων, η ανάγκη συμμετοχής τους στην οργανωμένη ε, κοινωνία των πολιτών, στο να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη, του ενεργού πολίτη, η απασχόληση, διάφορα ζητήματα δεν έχουν διαλάθει της προσοχής μας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι έγιναν κάποια σχόλια για τους δείκτες και για τα αποτελέσματα της στρατηγικής και θα ήθελα σε αυτό να απαντήσω. Αυτή τη στιγμή συντάσσουμε μια έκθεση για τους νέους που θα δημοσιευθεί όταν δημοσιεύσουμε την πρότασή μας για την ανανέωση της στρατηγικής μέσα στην Άνοιξη και εκεί θα έχουμε 41 δείκτες που θα μετρούν το πώς επηρεάζουν όλα αυτά τους νέους και Ταυτοχρόνως θα αξιολογήσουμε τη στρατηγική με τη βοήθεια των κρατομελών και ήδη μπορώ να πω ότι οι εκθέσεις των κρατών μελών είναι διαθέσιμες διαδικτυακά και αυτό μας δείχνει πώς, ε, ποια είναι η εμπειρία τους με την ε, ε, εφαρμογή της στρατηγικής. Χθες κάναμε μια, ε, πέρσι κάναμε την αξιολόγηση. Δεν θα σας, πω, δεν θα σας αναφέρω όλα τα ευρήματα, αλλά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Πέρσι είπαμε ότι ήταν η χρονιά της ακρόασης. Με, περιμέναμε τους δείκτες, τις έρευνες, αλλά και τις προσδοκίες των εμπλεκομένων. Περάσαμε αρκετό χρόνο ε, συζητώντας πέρσι Είχαμε την διάσκεψη των νέων στις Βρυξέλλες τον Μάιο και είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα και με χαρά θα σας τα ξαναστείλουμε και θα, σας τα, θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Υπάρχει το φόρουμ για τον, τους νέους και οι εκπρόσωποι των νέων αποφάσισαν να το διαρθρωμένο διάλογο με τους ε, ηθήνοντες να τον αφιερώσουν ε, στο θέμα του ε, μέλλοντος και της μελλοντικής στρατηγικής και θα σας ενημερώνω για την έκβαση αυτής της συζήτησης. Πολλά δηλαδή έχουν αρχίσει να προκύπτουν ως στοιχεία, ως πορίσματα. Ε, υπάρχει δηλαδή υλικό το οποίο είναι χρήσιμο για να αξιολογήσουμε πού έχει επιδράσει θετικά η στρατηγική και τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Σίλβια Κώστα και σύντομα. Ε, ναι, δεν είχα ακριβώ το λόγο, αλλά με χαρά θα πω ότι χαίρομαι για τι προτάσει τη ηγήτρια. Τι συμμερίζομαι απολύτω. Έχουμε να κάνουμε μια στρατηγική στιγμή, το είπε και η Επιτροπή νωρίτερα. Είμαστε μεταξύ τη διάσκεψη του 17 για την πολιτική για του νέου, ε, την ακρόαση για την οποία έγινε λόγο και τις νέες προοπτικές για, τη στρατηγική, για τη νέα στρατηγική για τους νέους. Ε, έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού που είναι πολύ μεγάλη επικαιρότητα γιατί δίνει στην κατάλληλη στιγμή κατευθύνσεις. Και μάλιστα πριν από το πολιτισμικο οικονομικό πλαίσιο ε, θα έχω να προτείνω λοιπόν τα εξή περισσότερο να προβάλλουμε τις οργανώσεις των νέων, τις, ε, τους συλλόγους ενός προσώπων λοιπά, Σε τοπικό ή άλλο επίπεδο που ενισχύουν και το ρόλο τους ως πολιτών αλλά και την ε, μόρφωση του, το μορφωτικό τους υπόβαθρο. Δεύτερον, από το Youth Forum προκύπτει το αίτημα για μια ομάδα εργασίας ε, διοργανικού συντονισμού, πέραν του διαρθρωμένου δηλαδή διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε αυτήν την προσέγγιση, την διατομεακή, πολιτικών, εκ των οποίων μάλιστα και ορισμένοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια πραγματική πλατφόρμα με κριτήρια αξιολόγησης ε, εξάντε και έξω. Κάποια κράτη μάλλον, μάλιστα το έχουν κάνει όπως η Αυστρία που έχει αρχίσει να δοκιμάσει το σύστημα της ε, αξιολόγησης λοιπόν των πολιτικών τρίτων και δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και για την εργασία βεβαίως αλλά για μας ως Επιτροπής ε, Πολιτισμού είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στη, στα ζητήματα των νίτς, των νέων που δεν είναι ούτε σε εκπαίδευση, ούτε σε κατάρτιση, ούτε σε επασχόληση και βέβαια άλλες διαστάσεις που ξεπερνούν τις απλές δεξιότητες, δηλαδή την πορεία της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, την, τη γραμμική αυτή δηλαδή προσέγγιση. Εμείς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μια προοπτική που θα δίνει και τη συνέχεια της ε, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ε, διαδικασίας. Επίσης έχουμε τη Σύνοδο του Γκότεμπορκ. Τελειώνω. Που, είναι, που δηλώνει ότι είναι πρωταρχική και κύρια διάσταση αυτή της εκπαίδευσης. Και έχουμε και μια σημαντική έκθεση της ΟΚΕ από τα συνδικάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει στοιχεία για την σημασία που μπορούν να διαδραματίσουν, που μπορούν να έχουν οι νέοι, οι προερχόμενοι από τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες, για να συμπληρώσουν αυτό το οποίο δεν προσφέρεται σε επίπεδο νέων ευρωπαϊκής καταγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Σε τρία λεπτά μπορείς να προσπαθήσει να μας ε, κάνεις τα συμπεράσματα. Ναι, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Γιατί ε, πολλά τα είπε η Σίλβια ούτως ή άλλως. Δεν μπορούμε να κατατμήσουμε αναηλικίες. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτή την εκπαιδευτική και κοινωνική διαδικασία. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπει το Child Guarantee, η εγγύηση για την παιδική ηλικία. Είναι μία από τις βάσεις έτσι ώστε η πολιτική για την νεολαία να μπορέσει να αναπτυχθεί. Το σχόλιο του κυρίου Μαρίνου ήταν πολύ ε, ενδιαφέρον. Κύριε Μαλινόφ, έχετε δίκιο. Μέρος της νεολαίας συμμετέχει στις οργανώσεις των νέων και θέλει να είναι ενεργός πολίτης, άλλοι όχι και πρέπει αυτούς να ενθαρρύνουμε και να τους διευκολύνουμε στη συμμετοχή τους. Άλλο κομμάτι όμως της νεολαίας δεν νιώθει καθόλου έτσι και πρέπει να δουλέψουμε όντως, να το τονίσουμε αυτό, να καταφέρουμε Βεβαίως δεν είναι μόνο οι νέοι, κάποιοι νέοι, αλλά και σε άλλες ηλικιακέ ομάδες ε, πολλοί δεν αισθάνονται την ανάγκη να εμπλακούν. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε οι νέοι που το βιώνουν να αποκτήσουν ευρωπαϊκή συνείδηση και να συνειδητοποιήσουν γιατί είναι πράγματι τόσο σημαντικό η ενεργή ιδιότητα, ο ενεργός πολίτης. Δεν είναι ότι νιώθουν απαραίτητα αποκλεισμένοι, αλλά δεν νιώθουν αυτή την ανάγκη να συνεισφέρουν. Ζουν την ζωή τους ησύχω και δεν εμπλέκονται. Αυτό ε, πρέπει να το καλλιεργήσουμε, δηλαδή την αντίθετη τακτική και επιθυμία και θα υπάρξουν προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές ομάδες τις οποίες ως εισηγήτρια θα προσπαθήσω να συγκεράσω. Το σημαντικό είναι να βασιστούμε ε, στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στις οργανώσεις των νέων θα έχουμε πολλές συνεδριάσεις και με τις οργανώσεις των νέων παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης και μεγάλο μέρος της ανάλυσης της στρατηγικής προήλθε από τις οργανώσεις των νέων και η Κομισιόν μπορεί να το βεβαιώσει αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστώ πολύ και πολύ καλή επιτυχία στην προσεχή δουλειά σα. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση. Και νομίζω δίνει και ενδείξει για το τι μπορούμε να περιμένουμε για, από μια μελλοντική στρατηγική για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 Μαρτίου 11 κνέει προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 25 Απριλίου. Έκθεση ελπίζουμε ότι θα πάει το Μάιο στην Ολομέλεια και Προχωρούμε. Στο επόμενο θέμα. Γνωμοδότηση έκθεση πρωτοβουλίας. Έβδομη έκθεση για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας, εδαφικής συνεργασίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός. Ο συνάδελφος κύριος Διάκον, Διάκονο έχει το λόγο ως εισηγητής παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ίσως η μαγική λέξη διάλειμμα να προφερθεί κάποια στιγμή. και είχα υποβάλει προτάσεις για τη χρηματοδότηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, τους τελευταίους δύο κύκλους του προϋπολογισμού και η απάντηση της Επιτροπής ήρθε μετά την σύνταξη της γνωμοδότησης, άρα θα πρέπει να τη συμπεριλάβω ως τροπολογία, ως προς το συνολικό ε, ποσό το οποίο ανέρχεται στα 11 δις ευρώ. 11 δις ευρώ λοιπόν είναι ένα καθόλου αμεληταίο ποσό. Το σημαντικό όμως είναι προς τα πού πηγαίνουν τα χρήματα. Είχαμε πολλά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, καλές επενδύσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία που οδήγησαν στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, ολόκληρων περιφερειών. Δυστυχώς όμως έχουμε και κακά παραδείγματα που οδηγησαν στην αναπτυξη ολόκληρη της περιοχης ολοκληρων περιφερειων δυστυχως ομως εχουμε και κακα παραδειγματα που οδηγησαν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μνημεία που επισκευάστηκαν ή αναστηλώθηκαν με άσχημο τρόπο ή που τελικά έμειναν ερήπια και δεν αναστηλώθηκαν και δεν αναπαλαιώθηκαν. Ε, σε όλες τις συζητήσεις για το έθος της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, προκύπτει ε, ξανά και ξανά η διαπίστωση ότι χρειαζόμαστε σωστή επένδυση και σωστή αξιολόγηση καθ' όλη τη διάρκεια του εκάστοτε προγράμματος. Άρα και σωστές στρατηγικές, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, ώστε οι επενδύσεις να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια. Να μην ξεχνάμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην οικονομία. Στην οικονομία. Οι μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν σαφέστατα αποδείξει ότι δεν είναι έργα φιλανθρωπίας οι επενδύσεις αυτές, δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη, ε, ενισχύουν το εμπόριο, τον τουρισμό. Ε, υπάρχει ένας κύκλος δηλαδή εξωτερικός δραστηριοτήτων πολύ σημαντικός. Με ενδιαφέρον είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρει ποτέ τον πολιτισμό στην 7η έκθεση. Ελπίζω όμως όλες αυτές οι πτυχές που αναφέρω εδώ να ληφθούν υπόψη. Στην επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στηρίζομαι στην υποστήριξή σας. Να μην αφήσετε την εκπαίδευση και τον πολιτισμό να είναι ένα δευτερογενές ε, κομμάτι της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διάκονου και ξεκινούμε με τους ε, σκιώδεις. Ο Μπογκδάν Βέντα έχει το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του. Συμφωνώ μαζί του. Η εκπαίδευση και ο αθλητισμός έχουν μεγάλες δυνατότητες ως προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ως προς τη συμβολή τους στην ε, ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει και αυτοί οι τομείς πολιτικής να συμπεριληφθούν. Έχουμε για παράδειγμα το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ε, τα διαρθρωτικά ταμεία ε, που μπορούν να συμβάλλουν και στα ζητήματα της ε, νεολαίας. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστούν όλα αυτά μέσω του Ταμείου Συνοχής. Οι περιφέρειες έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό ε, στα κλάστερ και στην δημιουργική βιομηχανία ε, και ε, υπάρχουν επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση που συμμετέχουν ενεργά, κέντρα που συμμετέχουν ενεργά, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί όλα τα στοιχεία και χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση ε, είναι βέβαιο ότι μπορεί η συμμετοχή να αυξηθεί. Ε, η πολιτική μας θα πρέπει να ενισχύσει μια τέτοια κατεύθυνση και με τη βοήθεια των ε, διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής. Έχω ένα ερώτημα. Αυτά τα στοιχεία που ε, συμπεριλαμβάνονται στην γνωμοδότησή σας, ποιες χρονιές, ποια έτη αφορούν. Εγώ βεβαίως ε, θα ε, υποβάλλω και τροπολογίες και προσβλέπω στην καλή συνεργασία που θα έχουμε με τον κύριο Τιακονού. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίλβια Κώστα έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω τον εισηγητή. Είχαμε μια σημαντική και ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση ως σκιώδης. Βεβαίως θεωρώ ότι πρέπει να σωματώσουμε τα εξή θέματα. Είναι πολύ σοβαρό το γεγονό δεν υπάρχει καμία αναφορά στην έκθεση τη ε, επιτροπή για την Οικονομική Συνοχή στην 7η έκθεση. Δεν υπάρχει αναφορά στον πολιτισμό. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είχαμε προτείνει, η συνάντηση δηλαδή τη Επιτροπής Πολιτισμού με την Περιφερειακή, ίσως και μια ακρόαση, να καλέσουμε δηλαδή σε ακρόαση τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών, ε, Περιφερειακής Πολιτικής θα είναι πολύ δύσκολο να συστήσουμε διδάλω τα θέματα στην ουσία τους. Ένα άλλο θέμα είναι σημαντικό πιστεύω στον προγραμματισμό μας να ορίσουμε συγκεκριμένα και ειδικά θέματα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Ξέρουν οι συνάδελφοι ότι ο πολιτισμός ενσωματώθηκε μετά τους ε, περιβαλλοντικούς, ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς και τους πολιτιστικούς ε, θησαυρούς όρος πολιτισμός. Επομένως, ο όρος, η διάσταση ε, του αστικού κέντρου, η διάσταση της υπαίθρου ή ως συνδυασμένη διάσταση χωροταξική του πολιτισμού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να μιλήσουμε και για επενδύσεις στη γνώση, στις νέες δεξιότητες που ε, υπηρετούν την ε, διαχείριση του πολιτιστικού προϊόντος ποιότητας. Εδώ δεν υπάρχουν δείκτες, το ζητούμε εδώ και καιρό, για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των περιφερειακών πολιτικών για τον πολιτισμό, μεγάλο έλλειμμα πιστεύω, είναι σημαντικό ως Επιτροπή Πολιτισμού να επεξεργαστούμε προδιαγραφές ποιότητας για την αξιολόγηση, για τη διαχείριση του πολιτισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως έχουμε και στην έκθεσή σου ζητήσει. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι επενδύσεις στο ψηφιακή τεχνολογία, στο ευρύ φάσμα στο και στο ε, άκρος ευρύ φάσμα και όλο το υπόλοιπο αυτό σύστημα υποδομών τεχνικών και μη αφορά και τα μουσεία και όλους τους θεματοφύλακες πολιτιστικού υλικού Πρέπει επομένω να προαχθεί στο πλαίσιο των σημαντικών παρεμβάσεων σε υποδομές που χρηματοδοτούνται με τον κανονισμό της συνοχής. Ευχαριστώ. Κύριε Εύανς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή Λίγα σχόλια έχω να κάνω. Καταρχάς το σημείο 4 είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ρητή αναφορά στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η συνοχή για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη σημασία του πολιτισμού, της κουλτούρας και της εκπαίδευσης δεν γίνεται να υπερβάλλουμε. Όσε φορές και να το λέμε, υπερβολή δεν είναι. Γιατί έτσι αναπτύσσεται το άτομο, αποκτά την ταυτότητά του και συμβάλλει στην κοινωνία, ε, συμβάλλει στην οικονομία και δημιουργεί μια πιο συνεκτική κοινωνία. Δεν, ε, η ισότητα είναι το ε, εκ των ουκάνευ. Άρα πρέπει να μπορέσουμε να μετρούμε την, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τη συμβολή του, την εκπαίδευση, τη σχέση μεταξύ αυτών για να επιλέγουμε και τα καλύτερα έργα και προγράμματα. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή μου πώς θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ε, ενδιαφέρουσες συνεισφορές. Καταλαβαίνουμε καλύτερα και προετοιμαζόμαστε καλύτερα έτσι για τις επόμενες εκθέσεις που θα συντάξουμε και θα δημοσιεύσουμε. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι βεβαίως ε, μπορούμε να βελτιωθούμε. Θα πρέπει να κάνουμε καλύτερες εκθέσεις. Να σας επενθυμίσω περί τίνος πρόκειται. Η έκθεση για τη συνοχή ε, τη συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει ένα στιγμιότυπο για το πώς αποδίδουν οι περιφέρειες, ποιες είναι οι επιδόσεις τους. Δεν δίνουμε... Ε, δεν λέμε τι έχει γίνει με την πολιτική συνοχή, ποια ήταν η χρηματοδότηση, ποιες ήταν οι παρεμβάσεις και το καθεξής. Στις εκθέσεις αξιολόγησης ο πολιτισμός Ε, έχει πολύ μεγαλύτερο μέρος αφιερωμένο σε αυτόν από ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά για να καταλάβετε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Η έκθεση ασχολείται πολύ περισσότερο με την εκπαίδευση, την αναγνωρίζει ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την ανάπτυξη των περιφερειών και σίγουρα θα δείτε ότι πολλά από τα στοιχεία είναι εκεί, βρίσκονται για να μας δώσουν ένα στιγμιότυπο για τις επιδόσεις των περιφερειών στον τομέα της εκπαίδευσης. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με τον πολιτισμό, γιατί υπάρχει έλλειψη δεδομένων και στοιχείων. Αν είχαμε δεδομένα και στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο, με χαρά θα συμπεριλαμβάναμε περισσότερα κείμενα και εδάφια για τον πολιτισμό στην έκθεση. Άρα να ασκήσουμε λόμπι, να χρησιμοποιήσουμε συνέργειες, να συνεργαστούμε για να αποκτήσουμε περισσότερα στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο για να μπορέσουμε να τα αποτιμήσουμε, να τα αξιολογήσουμε, να τα μελετήσουμε και άρα να τα περιλάβουμε στην πρότασή μας και στην εκθεσή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όταν όμως υπάρχουν δεδομένα θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να καλούνται να τα παραδίδουν ώστε να μπορούν και να αξιοποιούνται τα στοιχεία αυτά. Ίσως αυτό θα ήταν ένα πρώτο καλό θετικό βήμα, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια συνολικότερη εικόνα. Κύριε Διακονού, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, τα κύριε Βέντα, τα 11 δις έχουν να κάνουν με τον ε, κύκλο του προϋπολογισμού μέχρι το 2020. Περιμένουμε απαντήσεις και από τα Υπουργεία και από, τις, ε, από την Επιτροπή και θα σας τα στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κυρία Κώστα, αλλά και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στρέφουμε προς εσάς για να πω ότι έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά επανειλημμένως με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέσαμε ερωτήματα όπου μπορούσαμε και μία από τις πιο καταπληκτικές απαντήσεις και χαίρομαι που έχει υπάρξει πρόοδος έκτοτε ήταν η εξής που ε, απάντηση που πραγματικά μας κατάπληξε. Αναφέρουν τον πολιτισμό στην αρχή, αλλά μετά το ξέχασαν στην έκθεση, όσο προχωρούσε η έκθεση, και όταν την ξαναείδαν είπαν δεν πειράζει, δεν θα το παρατηρήσει κανείς. Ίσως αυτό ήταν λάθος και ατύχημα, γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια απάντηση πολύ πιο ελπιδοφόρα για το μέλλον. Τώρα, το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες εδώ στην Επιτροπή ΚΑΛΤ, πολιτισμού δηλαδή, και όλοι μας πρέπει να προσεγγίσουμε τον πολιτισμό ως μέρος της εκπαίδευσης, γιατί είναι ένα ανώτερο τμήμα της εκπαίδευσης, δεν μπορούμε να το δούμε αλλιώ. Άρα, είναι απαραίτητο αυτός ο τομέας, η, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, να, ε, αυτές οι συνιστώσεις του πολιτισμού να συνεργάζονται και να ε, μπει αυτό και στις πολιτικές ομιλίες και στις ε, πολιτικές γενικότερα να μην είναι κενά λόγια, αλλά θεμελιώδης πτυχή, κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη, για την ε, καλλιέργεια του, της αίσθηση του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Χωρίς κουλτούρα και χωρίς πολιτισμό δεν έχουμε και τίποτα ως Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διάκονο. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 27 Φεβρουαρίου, 2 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Μαρτίου και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης που θα συζητηθεί και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό και θα παρακαλέσω όλους όσοι δεν είναι ευρωβουλευτές ή δεν εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκαταλείψουν την αίθουσα το σύντομότερο δυνατό και όσο γίνεται πιο ήσυχα.